για την ισότητα των φίλων και τα δικαιώματα γυναικών και ανδρών μετά το 2015. Δίνω τον λόγο σε μία εκ των συντακτών, την κυρία Γκαρθία Πέρες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά, Μιλούμε για ισότητα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σίγουρα, πολλοί από τους παρόντες και τις παρούσες σε αυτή τη συζήτηση θα ήθελαν να καθίσουν και να ακούσουν όλα αυτά που έχουμε να πούμε. Γιατί η ισότητα είναι πραγματικά προτεραιότητα και στη δική μας δουλειά και στη δική μας πολιτική ιδεολογία. Οι γυναίκες είναι το 50% του πληθυσμού στην Ευρώπη και δεν μπορείτε εσείς να ασκείτε πολιτική σε δικό μας βάρος. Επομένως το πρώτο που ζητούμε είναι να μας ακούσετε εσείς πολιτικοί άνδρες και να γνωρίζετε πολύ καλά ε, τις ερωτήσεις που απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δρομολογήσει πολιτικές ισότητες μεταξύ γυναικών και ανδρών. Γιατί μιλούμε για μια αξία, για μια αρχή θεμελιώ, ε, εγχείρημα. Η ισχύουσα στρατηγική ολοκληρώθηκε το 2015. Τον Ιούνιο του 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε συγκεκριμένη θέση στη συζήτηση για το ποιο περιεχόμενο θα πρέπει να είναι και ποιες θα πρέπει να είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που θα πρέπει να περιλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη νέα τη στρατηγική για τα θέματα των φύλων, των δύο φύλων και την ισότητα ανδρών και γυναικών. Και έγινε δημόσια διαβούλευση και το 90% και πέρα των ατόμων που ε, συμμετείχαν στη δημόσια διαβούλευση τάχθηκαν υπέρ του επίγοντος χαρακτήρα. Είναι απαραίτητο η πολιτική προτεραιότητα να μεταφραστεί σε δέσμευση, συγκεκριμένη δέσμευση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιτροπή πρέπει να ανακοινώσει νέα στρατηγική για το θέμα αυτό. Από τον Ιούνιο του 2015 που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε συγκεκριμένη θέση και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει αυτή τη δουλειά, από τότε περιμένουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και πώς απάντησε η Επιτροπή. Το Δεκέμβριο του 2015 υιοθέτησε ένα έγγραφο εργασίας που συνέταξαν οι αρμόδιες της υπηρεσίες ένα έγγραφο το οποίο είναι απολύτως σεβαστό, είναι ένα περιεχόμενο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, όμως δεν περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη δέσμευση, πολιτική δέσμευση που θα πρέπει να υπάρχει. Ένα έγγραφο εργασίας δεν έχει προϋπολογισμό. Ένα έγγραφο εργασίας δεν παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν τα προτινόμενα μέτρα. Ένα έγγραφο εργασίας δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Όμως για να εφαρμοστούν οι πολιτικές πρέπει να έχουμε προεπολογισμό και μηχανισμούς αξιολόγησης. Επομένως ένα έγγραφο εργασίας δεν είναι γι' αυτό το λόγο δέσμευση, πολιτική δέσμευση. Επιμένουμε να υιοθετηθεί συγκεκριμένη στρατηγική για την ισότητα των δύο φύλων α, και να υιοθετηθεί αυτή η στρατηγική από το Σώμα των Επιτρόπων γιατί πρέπει να είναι πολιτική δέσμευση του συνόλου ε, του Σώματος των Επιτρόπων. Οι Επίτροποι όλοι πρέπει να το συζητήσουν και να το εγκρίνουν. Την πολιτική δηλαδή ε, ε, ισότητα των φύλων γιατί μιλούμε για μισθολογικό χάσμα, Μιλούμε για βία ε, ενδοοικογενειακή ή βία που ασκείται σε βάρος των γυναικών. Μιλούμε για ζητήματα θεμελιώδη στην πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε ικανοί να δρομολογήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Τα τελευταία χρόνια, εκτός από τις διάφορες κρίσεις που έχουν σημειωθεί στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, την οικονομική κρίση, την προσφυγική κρίση, την κοινωνική κρίση, εκτός από όλα αυτά και πέρα από όλα αυτά, αυτοί που υποφέρουν περισσότερο από όλες αυτές τις κρίσεις είναι οι γυναίκες. Θα πρέπει η διάσταση του φύλου να είναι ενσωματωμένη σε όλες τις πολιτικές, να είναι οριζόντια παρόν το θέμα αυτό σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα συνεχίσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεκδικούμε. Θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτή την ευκαιρία ε, για να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει γιατί δεν υιοθέτησε νέα ανακοίνωση δημοσίως και με διαφανή τρόπο ανακοίνωση για τη στρατηγική της για την ισότητα ε, των φύλων. Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν ενέκρινε ένα τέτοιο είδου έγγραφο δεν το συζήτησε ε, και δεν το υιοθέτησε ως σώμα επιτρόπων. Και γιατί πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να συζητήσετε πώς μπορείτε να προχωρήσετε τα θέματα ισότητα σε κάθε μία από τις γενικές διευθύνσεις, σε κάθε ένα από τα διαφορετικά χαρτοφυλάκια των διαφορών Ευρωπαίων επιτρόπων και να μας πείτε πώς θα συνεργαστείτε με το τρίο ε, των Προεδριών του Συμβουλίου έτσι ώστε να υπάρξει στρατηγική ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είτε θεμελιώδες και είναι απαιτητό. Θα θέλαμε να ήταν εδώ η κυρία Γιούροβα, η αρμόδια επίτροπος ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως δεν είναι επιμέρους πολιτική η πολιτική της ισότητας των φύλων. Είναι μια πολιτική εγκάρσια, οριζόντια ε, και η δέσμευση της Επιτροπής πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Και τώρα εξ ονόματος ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ανδρουκάητης. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να ξεκαθαρίσω τις προθέσεις τη Κομισιόν για την πολιτική της ισότητας ε, στη διάρκεια της ε, θητείας μας. Η Κομισιόν δημοσίευσε την ε, στρατηγική της για το φύλλο 2016-2019 στι 3 Δεκεμβρίου του 2015 ως πλαίσιο για μελλοντικές δράσει για να βελτιωθεί η ισότητα των φύλων. Η στρατηγική αυτή είναι συνέχεια της στρατηγικής ε, της ε, Κομισιόν για ισότητα μεταξύ των δύο φύλων 2010-2015. Η στρατηγική, οι προτεραιότητε της στρατηγικής εξακολουθούν να ισχύουν. Η διαβούλευση και η αξιολόγηση που κάναμε για να προετοιμάσουμε την στρατηγική μας αυτή, το επιβεβαιώνουν. Ενώ έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, απαιτείται περαιτέρω δράση για να επιτύχουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Η ισότητα των φίλων είναι σημαντικό κομμάτι της, ε, του προγράμματος της Κομισιόν Γιούνκερ. Όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε και ένα πρόγραμμα καλύτερης νομοθεσίας, επανασχεδιάζοντας τις δραστηριότητες και τα μέσα μας. Ως Επίτροπος μπορώ να σας επιβεβαιώσω πως η νέα στρατηγική δέσμευση είναι η νέα μας πολιτική και έχει την πολιτική στήριξη ολόκληρης της Κομισιόν. Παρουσιάζεται επίσης το πρόγραμμα εργασίας του 2016. Καταβάλουμε πρακτικές προσπάθειες για να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων, όπως εξηγήθηκε σε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Γυναικών τον Δεκέμβριο πρέπει να εστιάσουμε στα αποτελέσματα στο έδαφος. Περιγράφουμε λοιπόν στην δέσμευσή μας το πώς θα εστιάσουμε σε πέντε τομείς προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της εντολής μας. Στο να αυξήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, να μειώσουμε το χάσμα πληρωμών και συντάξεων και να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια των γυναικών, να προωθήσουμε την ισότητα ανδρών και γυναικών στη λήψη αποφάσεων, να καταπολεμήσουμε την βία με βάση το φύλλο, να προωθήσουμε τα δικαιώματα των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης, επιβεβαιώνουμε την ένταξη αυτής της πολιτικής σε όλες τις πτυχές των παρεμβάσεων της Υπάρχουν πάνω από 30 δράσεις κλειδιά που θα εφαρμοστούν στους πέντε τομείς προτεραιότητας που ανέφερα. Πέρα από στόχους και χρονοδιαγράμματα. Επίσης θα δούμε ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης ταυτόχρονα με την ανάπτυξη δικτών έτσι ώστε να έχουμε μια ένα μέτρο σύγκρισης με βάση το οποίο θα αξιολογήσουμε την πρόοδο. Η στρατηγική μας αυτή δέσμευση βασίζεται στους στόχους που έχουμε συμφωνήσει στο επίπεδο της Ένεσης. Συγκεκριμένα στηρίζει το να επιτύχουμε τους στόχους του 2020 για 75% ποσοστό απασχόλησης άνδρων και γυναικών. Ένα συγκεκριμένο μέσο προγραμματισμού για την Κομισιόν, στο οποίο ευχαρίστω μπορούν να εμπλακούν και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Στις 15 Ιανουαρίου η Κομισιόν συμμετείχε σε ομάδα εργασία του Συμβουλίου για κοινωνικά ζητήματα, όπου έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την στρατηγική μα δέσμευση. Η Ολλανδική Προεδρία εξέφρασε την πρόθεσή της να εγκριθούν συμπεράσματα του Συμβουλίου στην συνεδρίαση του Μαρτίου. Η στρατηγική αυτή δέσμευση αποτελεί μια βάση για τις δράσεις ισότητας των φύλων τα επόμενα χρόνια, ε, ιδιαίτερα καθώς καλύπτει τα βασικά ζητήματα που αναγνώρισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο στο ψήφισμα του Ιουνίου 2015. Είναι το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν για το 2016 μέχρι 2019. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ε, Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σα ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα θα ακούσουμε τις εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων για το ΕΛΚ η κυρία Κωνσταντς Λεγκρίπ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ στο ημικύκλιο του Κοινοβουλίου του Στρασβούργου για να συζητήσουμε εκ νέου το κρίσιμο θέμα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, με βάση μια προφορική ερώτηση που ορισμένες πολιτικές ομάδες θέλησαν να απευθύνουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που στιγμάτιζε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δημοσιεύσει έγγραφο για ένα συγκεκριμένο είδος καθεστώτος, μια ανακοίνωση ή στρατηγική ανακοίνωση, αλλά δημοσίευσε για, ως ε, οδικό χάρτη για να υπογραμμίσει τις δράσεις της για την περίοδο 2015 μέχρι 2019, απλά ένα έγγραφο εργασία. Ειλικρινά, προσωπικά, και εξ του ΕΛΚΑ δεν με ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλες αυτές οι συζητήσεις ε, του περί καθεστώτος του ενός ε, ή του άλλου εγγράφου. Αυτό που έχει σημασία είναι η πολιτική, ο δυναμισμός, ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζονται οι δράσεις αλλά και οι διαδικασίες, η μεθοδολογία. Μέσα σε αυτή την προοπτική, η μεθοδολογία, οι τομεί δράση και οι δεσμεύσει που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επίτροπο Γιούροβα στο έγγραφο εργασία αντιστοιχούν ακριβώ στι προτεραιότητε τις ανησυχίες ε, του ΕΛΚ. Θέλουμε συγκεκριμένη ρεαλιστική και αποτελεσματική προσέγγιση. Ε, συγκεκριμένους ε, μετρήσιμους στόχους, διαδικασίες αξιολόγησης, να τονίσουμε την ανάγκη να μεταγράφονται σωστά και να εφαρμόζονται σωστά οι φυστάμενε νομοθεσίες πριν να προβλέψουμε ενδεχόμενε νέες νομοθετικές προτάσεις, εν ολίγης να είμαστε χρήσιμοι, συγκεκριμένοι και ρεαλιστές και να επικεντρώσουμε σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως χρήσιμο στο ευρωπαϊκό ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο να πιέσουμε τα κατημέλη ώστε να αντιμετωπίσουν τις ευθύνες τους και να τις αναλάβουν. Αυτή η πολιτική βούληση σαφώς είναι γεγραμμένη στο πρόταση ψηφίσματος του ΕΛΚΑ και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, εξ ονόματος των σοσιαλιστών, η κυρία Νόχλα. Αγαπητοί συναδελφοί, εμείς είμαστε οι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού λαού. Εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς η πλειοψηφία των βουλευτών απαιτούμε σήμερα εκ νέου τα δικαιώματά μας. Έχουμε μοραλή. Ηθικό δικαίωμα στο να προωθηθεί η ισότητα. Και έχουμε βεβαίως και μεγάλη αυτοπεποίθηση. Έχουμε ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ζητάει από την Κομισιόν να προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα. Ομόφωνα επίσης έχουμε την στήριξη των κρατών μελών που στηρίζουν αυτή τη στρατηγική και έχουμε την στήριξη των πολιτών της Ένωσης που στο πλαίσιο δημοσκοπήσεων τάχθηκαν κατά πλειοψηφία υπέρ της ισότητας. Συνεχώς, η κυρία Γιώροβα λυπάται για το ότι ε, και μας λέει μάλιστα ότι ένα εσωτερικό έγγραφο εργασίας είναι το ίδιο με μια στρατηγική, αλλά ξέρει ότι αυτό δεν ισχύει. Αυτό το οποίο μας ε, υπέβαλε είναι ένα χλιαρό έγγραφο και άρα πρόκειται για υποβάθμιση του θέματος της ισότητας και των ανθρώπων στην Ευρώπη. Σήμερα προσωπικά μίλησα με τον Μάρτιν Σούλτς και επεσήμανα αυτό το θέμα. Θα έρθει σε επαφή με τον κύριο Γιούνκερ για να ζητήσει δικαιοσύνη για το κοινοβούλιο, γιατί το αξίζει αυτό το κοινοβούλιο. Όποιος είναι κατά των δικαιωμάτων των γυναικών εξασθενεί την Ευρώπη. Όποιος είναι κατά της ισότητας είναι σεξιστής. Όποιος εμποδίζει μια στρατηγική παραβιάζει δημοκρατικές αρχές. Θέλουμε μια στρατηγική και τη θέλουμε τώρα. Έχουν υποθεί τα πάντα. Τα 30 δευτερόλεπτα που μου απομένουν θα ήθελα να τα δώσω στην κυρία Γιώργα για να σκεφτεί. Ε, έχω, έχω χρόνο ομιλίες ακόμα. Όχι, όχι, έχω 10 δευτερόλεπτα. Ελπίζω να σκεφτήκατε και η κυρία Γιώροβα και εσείς και να έχουμε τελικά στρατηγική. Ευχαριστώ. Ε, on behalf ε, ECR e, e, Εξ ονόματος του ECR, η κυρία Βυσνιεύσκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπα, αξιότιμοι συνάδελφοι. Η αριστερά θέλει να προωθήσει ιδεολογικά τα θέματα του φίλου ε, για να κάνει τα παιδιά σεξουαλικά όντα, να προωθήσει τις ε, ε, LGBTI και να Καταλήξουμε τελικά σε μια κοινωνία όπου η παραδοσιακή οικογένεια μπορεί να θεωρεί ότι υπόκειται διακρίσει γιατί δεν είναι αρκετά σύγχρονη, δεν είναι αρκετά ευρωπαϊκή, γιατί είναι, βάση περιπτώσει, ξεπερασμένη. Ο αριθμός των κανονισμών που υπάρχουν όσον αφορά τα μέτρα κατά των διακρίσεων είναι τεράστιος. Δεν χρειάζεται να υιοθετηθούν νέοι κανονισμοί. Η ομάδα μου είναι κατά των νέων ψηφισμάτων ε, της αριστεράς. Εμείς προτείνουμε μια διαφορετική και πιο λογική προσέγγιση. Είναι ο καιρό να επανέλθουμε στι ρίζε μα και να βασιστούμε στι αξίε ε, των οποίων οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην ντρεπόμαστε για τη χριστιανική μα κληρονομιά. Είναι αυτού του είδος η σοφία και η δύναμη που μας χρειάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μλίναρ. Για δύο λεπτά. Very much, Mr. President. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο Γιούροβα για τι προσπάθειε που κατεβάλλει ώστε να μετατραπεί σε πραγματικότητα η ισότητα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δείξει ότι είναι πραγματικά αφοσιωμένη και προσιλωμένη σε αυτό το θέμα και κάνει προσπάθειες για τι διαπραγματεύσει με τι γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια και στο γεγονό ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να, να, δώσει όθηση στη... στο φάκελο για την άδεια μητρότητα ε, σε μια προσπάθεια για εξισορρόπηση της εργασιακής με την προσωπική ζωή. Ωστόσο δεν μπορώ να κρύψω την απογοήτευσή μου όταν αντιμετωπίζω ένα έγγραφο εργασία αντί για μια σωστή και ολοκληρωμένη στρατηγική υπέρ της ισότητας των φύλων. Δεν επικρίνω τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο, αλλά καταγγέλω στο όνομα της ομάδας μας την υποβάθμιση αυτής της στρατηγικής, ιδιαίτερα καθώς έχει γίνει ενάντια στη σαφή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, από την, εφόσον η έκθεση Νόιχελο υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία και ενάντια σε σαφείς δηλώσεις 22 κρατών μελών. Επιπλέον, η αξιολόγηση της περασμένης στρατηγικής ε, κατέληξε σε μια συγκεκριμένη έκκληση για περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής προσέγγισης που υιοθετήθηκε το 2010 και όχι στην αποδυνάμωσή της. Υπό το φως αυτών όλων ε, θα έπρεπε η ε, Κομισιόν και ολόκληρο το όργανο συλλογικά να εξετάσουν ε, ε, κατά πόσο αυτή η ανισότητα ε, η οποία επηρεάζει πάνω από το μισό πληθυσμό της Ευρώπης να είναι από, υποδέστερο από την γραφειοκρατία και μετά όπως και ο Μιλήτρια πριν από μένα έδειξε δείχνει ότι το θέμα της ισότητας των φύλων δεν το λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Mlinar, <laughs> not της Γκουε τώρα. Η κυρία ε, Μπιέρκ. Σα ευχαριστώ πολύ. Το Ευρωκοινοβούλιο συστηματικά εργάζεται ε, υπέρ της ισότητας. Μια νέα έκθεση για την ισότητα θα ήταν ένα καλό παράδειγμα. Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η εργασία υπέρ της ισότητας έχει τελματωθεί στην Κομισιόν και στο Συμβούλιο. Η απουσία ισότητας αντιστοιχεί στην ε, ανισότητα. Οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στους πόρους, ούτε στην, ε, στις ανώτατες θέσεις. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας. Χρειάζεται ένα πολιτικό όραμα και συγκεκριμένα μέτρα υπέρ της ισότητας. Γι' αυτό το Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, ε, θα πρέπει να φτιάξουν μια πολιτική υπέρ της ισότητας. Εάν μπλοκάρεται η πρόοδος, ε, σημαίνει άσκηση κυριαρχίας και ε, δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε αιώνες ε, παραδοσιακής καταπίεσης των γυναικών. Όχι, ευχαριστούμε. Εμείς θα προωθήσουμε τη στρατηγική υπέρ της ισότητας ε, και έχει πια φτάσει στη στιγμή να έχουμε μια Ευρώπη πιο φεμινιστική. Σας ευχαριστώ. On behalf of Για τους πράσινους. Η κυρία Ρέντκε. 1,5 λεπτό. Αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η ισότητα ανδρών και γυναικών πρέπει να την εγγυόμαστε σε όλα τα πεδία. Είναι σαφές και σύντομο το μήνυμα του άρθρου 23 της Ευρωπαϊκής Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και είναι σαφές το καθήκον μας ως νομοθετών, ημών στο Κοινοβούλιο, ημών με ύψιλο στο Συμβούλιο. Πώς μπορούμε να έχουμε μια κοινωνία όπου θα προστατεύουμε ε, τις ε, εργαζόμενες μητέρες και τους εργαζόμενους πατέρες. Πώς μπορούμε να έχουμε μια κοινωνία όπου θα έχουμε γυναικείες φωνές στις, στα ανώτατα ε, αξιώματα της οικονομίας. Για να μην υπάρχει βία εναντίον των γυναικών χρειάζομαστε εμπιστοσύνη, πολιτική βουλήση αλλά και σαφή στρατηγική. Έχω εκλεγεί σε ένα νομοθετικό σώμα για να κάνω πολλά πράγματα. Αυτό είναι αληθές, αλλά κυρίως για να διορθώσω νομοθετικά κενά και κυρίως νομοθετικά κοινά σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλές επιδόσεις σε αυτό, πρέπει όμως να κάνει παραπάνω. Ε, η απόσυρση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας. Έχει ανασταλεί η εξέταση της οδηγίας για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Δηλαδή υπάρχει οπισθοχώρηση στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά και αυτό είναι απαράδεκτο. Ας ε, κάνουμε το παν για να είναι επιτυχημένη η παρούσα θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι οι δουλειέ ε, του 20ου αιώνα οι οποίες μένουν κρεμείς και δεν έχουν τελειώσει τον 21ο αιώνα και αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Ντανιέλα Αγιούτο από το EFTD. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμη Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πάντοτε βρισκόμαστε στη γιορτή του ψεύδους και της υποκρισίας. Μιλάμε για μανιφέστα, συνθήματα και στόχους ιδεολογικού τύπου, αλλά που πόρο απέχουν από την πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς οι γυναίκες και τα προβλήματα που είμαστε υποχρεωμένες να αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Ε, ευχόμαστε μια ισότητα των φύλων που όμως μένει πάντα στον τύπο και δεν ε, βρίσκει στήριγμα σε καμία ουσιαστική πολιτική. Μιλάμε για λύσεις που μειώνουν ε, την ανισότητα ανάμεσα στα φύλλα, ωραία λόγια, αλλά αυτό που έχουμε κάνει και γράψει μέχρι στιγμή έχει χρησιμεύσει σε κάτι. Η ζωή των Ευρωπαίων γυναικών βελτιώνεται από χρόνο σε χρόνο ή η χειροτερεύει. Σοβαρά φαινόμενα διάκριση και ανισότητα που τόσο έντονα εμεί καταδικάζουμε εξακολουθούν να εμφανίζονται παρά τι ρυθμίσει και μα τα λένε οι εφημερίδε, τα στοιχεία που συλλέγουμε και οι οικονομικέ αναλύσει. Έχουμε επίση διαπιστώσει του τελευταίου μήνε ε, μετά αυτή το τελμάτωση για την οδηγία οδηγία για την ε, άδεια μητρότητα, αλλά και για εκείνη με τι γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια. Οι γυναίκε, ωστόσο, στην Ευρώπη είναι όλο ένα και πιο μόνε, πιο φτωχέ και όλο ένα και βιάζονται περισσότερο. Φτάνει πια. Πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένε και στοχευμένε δράσει και γρήγορα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ανασαμπόρσκα είναι ένα μισή σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όταν μιλάμε για ισότητα ανδρών και γυναικών μιλάμε εμέσως και για την μητρότητα. Το μισθολογικό χάσμα και τις διαφορετικές συντάξεις, το χάσμα των συντάξεων. Αυτά δείχνουν πόσο υποκριτική είναι η κοινωνία μας. μητρότητα και το να μεγαλώνει κανείς τα παιδιά δεν το θεωρούμε εργασία. Οι γυναίκες τιμωρούνται οικονομικά είτε λόγω του μισολογικού χάσματος, ε, της μικρής ε, άδειας μητρότητας, είτε γιατί δεν αναγνωρίζουμε το σημασία που έχουν οι γυναίκες για την κοινωνία. Μιλάμε για ελευθερία επιλογής των γυναικών και τους ασκούμε πίεση να μπουν στην επίσημη οικονομία. Κομισιόν και το Κοινοβουλίο πρέπει να εστιάσουν στις αιτίες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι ορισμοί. Ισότητα των φίλων που λέτε δεν σημαίνει ισότητα άνδρων και γυναικών. Δεύτερον, να αναγνωριστεί η σημασία της μητρότητας και της φροντίδας που παρέχουν οι γυναίκες στις οικογένειες. Μόνο τότε θα έχει νόημα η συζήτησή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Ζαμπόλσκα. Με συγχωρείτε, η κυρία Μαρία Αρένα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Επίτροπε, γιατί η ισότητα γυναικών και ανδρών ως ε, θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αξίζει περισσότερα. Δεν αξίζει περισσότερα από μία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί δεν αξίζει ένα πραγματικό πρόγραμμα με ε, συγκεκριμένο προϋπολογισμό, με αξιολόγηση, με μέτρα διοικητικά, αν αυτό είναι απαραίτητο. Ζητώ συγγνώμη, αλλά υπάρχουν προβλήματα με το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών, παραμένουν οι διακρίσεις, παραμένει η βία, παραμένουν τα σεξιστικά στερεότυπα. Ξαναθέτω λοιπόν το ερώτημα, γιατί δεν υπάρχει ανακοίνωση ή και περισσότερα πράγματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα σωρό ανακοινώσει της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει βγάλει ανακοίνωση για το επίπεδο ήχων και ηχορύπανση των κινητήρων, για τα μη επαδρομένα αεροσκάφη, για, τα ταξιδιωτικά πακέτα ένα σωρό ανακοινώσεις έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί παντός επιστητού. Αλλά για το θέμα των γυναικών υπάρχει διοικητική απλούστευση και ριφίτ και αναστολή της, οδηγίας για, της εξέτασης της οδηγίας για την άδεια μητρότητας. Ε, ζητώ συγγνώμη κυρία Κωνσταντς ε, Λεγκρίπα, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό με τη σημειολογία όπως λέτε. Έχει άμεση σχέση με την πολιτική και σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ορίσει την ισότητα ε, των φύλων ως πολιτική της προτεραιότητα, δυστυχώς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλάμε για gender mainstreaming αναφερόμαστε στο άρθρο 8 Τη συνθήκη που λέει σε όλε τι δραστηριότητες η Ένωση θα προσπαθήσει να προωθήσει την ισότητα ανδρών και γυναικών. Δεν είναι δικό μου αυτό. Αυτό είναι απάντηση της Κομισιόν ε, στην ερώτησή μου για να ξεκαθαρίσει το τι εννοούμε gender στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το gender με βάση αυτό το οποίο λέει η κυρία Στρέλα Ροντρίγκε ε, και η λοιποί συνάλφοι δεν υφίσταται Μιλάμε για έναν τελείως λανθασμένο ορισμό. Gender δεν σημαίνει να διδάσκουμε στο δημοτικό σεξουαλική αγωγή ή να διδάσκουμε το πώς σκοτώνουμε μικρά παιδάκια. Ούτε σημαίνει σήμερα άντρας, αύριο γυναίκα ή κάτι άλλο. Σημαίνει πολύ απλά ισότητα ανδρών και γυναικών. Τελεία και παύλα. Όταν μιλάμε ισότητα πρέπει να μιλάμε και για το μέλλον. Και δεν υπάρχει καμία ισότητα όταν οι γονείς και οι άκληροι μπαίνουν σε ίδια μοίρα. Σας ευχαριστώ. Λουίς Μπούρς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Συμφωνώ με κάποιους από εσάς και αυτό είναι σπάνιο, γιατί πράγματι σημειώνω και εγώ την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το μόνο που έχει παράγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα έγγραφο εργασίας. Χρήσιμο. Εάν κανείς βρεθεί σε δημόσιο χώρο και πρέπει να πάει σε δημόσιες τουαλέτες και δεν υπάρχει εκεί χαρτί υγείας. Αλλά μάλλον άχρηστο σε οτιδήποτε άλλο. Νιώθω μεγαλύτερη δύναμη, νιώθω περισσότερη ασφάλεια ως γυναίκα με τη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όχι, το αντίθετο ισχύει. Πάρα πολλές γυναίκες στην κολονία, στη Σουηδία και αλλού νιώθουν το ίδιο με μένα. Τι νομίζετε ότι θα συνέβαινε όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τις πόρτες να έρθουν εκατομμύρια άνθρωποι από χώρες και από κουλτούρες που μεταχειρίζονται τις γυναίκες ως ε, πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τους ΛΟΑΔ ως ακόμα τρίτης ή τέταρτης κατηγορίας κατηγορίας. Στη κολονία και αλλού οι πολιτικοί, οι αρχές, ο τύπος πρέπει επιτέλους έδειξαν μάλλον ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για την πολιτική ορθότητα και λιγότερο για τα δικαιώματα των ε, γυναικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται την ύπαρξη τέτοιου είδους βίας και τι γίνεται και με τον τράφικιν. Η ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που εκμεταλλεύονται τα δίκτυα των εγκληματιών για να φέρνουν θύματα τράφικιν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό το δείχνουν πολύ συγκεκριμένες και σοβαρές έρευνες. Είναι το τέλειο περιβάλλον έτσι ώστε οι εγκληματικές συμμορίες να δρούν με ασυλία, με ατιμορρησία η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα αυτό είναι και θα συνεχίσει να είναι παταγώδης αποτυχία. Όσο παραμένει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες, η ΛΟΑΔ, όλη η κοινωνία είναι λιγότερο ασφαλής ε, και λιγότερο σίγουρη. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ. Η Τερέσα Χιμένεθ Μπεθερίλ Μπάριο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, λέμε τα ισπανικά αλλά νομίζω και σε άλλες γλώσσες ότι ένα δέντρο συχνά κρύβει το δάσος. Το σημαντικό σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι ο στόχος που έχουμε και ο τρόπος με τον οποίο θα τον πετύχουμε. Οι πιο προηγμένες κοινωνίες είναι οι κοινωνίες που έχουν σφυριλατήσει και προστατεύσει περισσότερο από τις άλλες τα δικαιώματα των γυναικών. Τον 20ο αιώνα πάρα πολλοί έχουν δώσει και, ακόμα και τη ζωή τους για να μπορούμε εμείς ως γυναίκες να καθόμαστε εδώ, να νομοθετούμε ε, για μια πιο δίκαιη κοινωνία τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε σε θέματα ισότητας είναι ψηλά. Το μισθολογικό χάσμα, για παράδειγμα, που είναι γραμμένο ότι μια γυναίκα πρέπει να κερδισει λιγότερο από έναν άνδρα για ε, δουλειά ίσης αξίας. Η βία ε, που έχει σχέση με το φύλλο. Ε, ένα σώρο νομοθετήματα έχουμε, αλλά πολύ μικρά και λίγα αποτελέσματα. Είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μεριμνήσει όλα αυτά να τηρούνται σε όλα τα κράτη-μέλη. Στηρίζουμε την πρακτική προσέγγιση που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη στρατηγική. Το σημαντικό είναι να μειωθούν οι ανισότητες. Αυτό πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Ξέρετε, οι γυναίκες δεν ενδιαφέρονται πώς θα ονομάσουμε την εκάστοτε στρατηγική. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να είναι αποτελεσματικές στρατηγικές και δεν πρέπει να μειώσουμε ούτε τους στόχους, να κατεβάσουμε τον πύχη των στόχων, αλλά ούτε να μειώσουμε και τα μέσα στη διάθεσή μας για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ευχαριστώ. Η κυρία Ροντρίγκες. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τα στοιχεία που έχουμε για την ισότητα των φύλων θα έπρεπε να μας οδηγήσουν να έχουμε μια συντονισμένη στρατηγική και αποτελεσματική για να καταπολεμήσουμε την ανισότητα και τις διακρίσεις. Από τα στοιχεία που έχουμε ήδη βλέπουμε πως χρειάζεται δράση, ε, οπότε είναι ακόμη πιο ανησυχητικά και εκείνα τα στοιχεία τα οποία μιλούν για την ανικανότητα της ε, Κομισιόν να συλλέξει ε, στοιχεία για την ανισότητα. Ας πούμε, ε, για την, ε, τον ακροτηριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων. Είναι γνωστό το τι συμβαίνει. Η Κομισιόν όμως δεν θέλει να δράσει. Τι γίνονται διαβουλεύσεις και άσχετες εργασίες διοργανικές φοβούμε ότι δεν έχετε καταλάβει καν γιατί ε, κάνουμε εμείς τέτοιου είδους ερωτήσεις. Μόνο έτσι μπορώ να συγχωρήσω αυτό το σχόλιο, την ιδέα δηλαδή της πολιτικής δράσης και της πολιτικής ενέργειας. Οι συνέπειες είναι, της, της μάλλον είναι πολύ σημαντικές και Εν τω μεταξύ πεθαίνουν περισσότερες γυναίκες. Μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα. Το 50% των... του πληθυσμού είναι δεύτερη δεύτερης κατηγορίας. Και αυτό αντικατοπτρίζει ακόμα κάτι. Την έλλειψη σεβασμού απέναντι στις γυναίκες. Η κυρία Γιούροβα λείπει σήμερα και αυτό το αποδεικνύει. Το ότι δεν έχει σεβασμό για τις γυναίκες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και ζητώ συγγνώμη για την κύρια Επίτροπο βρίσκεται σε άλλες διαπραγματεύσεις για την προστασία των δεδομένων και λυπάται για το ότι δεν μπορεί να ακούσει αυτή την συζήτηση. Το κείμενο είναι πρακτικό, χωρίς ιδεολογικές ε, μεγαλοστομίες. Σημαντικά για εμένα είναι η εφαρμογή και η παρακολούθηση. Αυτά για μένα μετράνε περισσότερο από τις υποσχέσεις. ε, λείπει εδώ πέρα το να αποτελέσει η Κομισιόν παράδειγμα και τα ηγετικά της τελέχη να είναι 40% γυναίκες. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους στόχους. Γυναίκες, ε, οι γυναίκες βεβαίως πρέπει να κάνουν παιδιά, να φροντίσουν και τους γέρους και ταυτόχρονα να δουλεύουν ε, όλες. Και τι κάνει η Κομισιόν. Η πρέπει να στηρίξει τις ευέλικτες μορφές εργασίας για να μπορούν και οι γυναίκες να δουλέψουν. Και εδώ πέρα πρέπει να κινητοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να εκτιμήσουμε περισσότερο τις ε, γυναίκες που θα ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Γιατί είναι το σημαντικό αυτό. Η, νομίζω η ομάδα η οποία εφίσταται τις περισσότερες διακρίσεις είναι οι γυναίκες που ασχολούνται με τα παιδιά και τους ε, γέρους και έτσι επενδύουν στο μέλλον της Ευρώπης και όχι ε, να, και δεν μπορούν να πληρώσουν για την δική τους σύνταξη. Αυτές πρέπει να στηρίξουμε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νταντσίλα έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παρουσίαση της στρατηγικής ε, της ισότητας ε, των δύο φίλων για το 2015 είναι κάτι το κατεπήγον ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό απαιτείται να γνωρίζουμε καλύτερα το πρόβλημα εις βάθος, να γνωρίζουμε τα, της αγοράς της εργασίας ε, και να προσαρμοστεί η νομοθεσία βεβαίως πρέπει να δούμε και την βελτίωση των δεξιοτήτων και της ε, ισότητας ε, και βεβαίω ε, και στον δημόσιο τομέα αλλά και στους κοινωνικούς εταίρους, στην κοινωνία των πολιτών και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και βεβαίως θα πρέπει να στηρίξουμε και τις γυναίκες επιχειρηματίες και τις δραστηριότητες των γυναικών οι γυναίκες ε, στην Ευρώπη αμείβονται με 17,8% λιγότερο από τους άντρες. Το μισθολογικό αυτό χάσμα έχει επιπτώσεις στη ζωή των γυναικών και στο εισόδημά τους αλλά και στις συντάξεις. Αυτόχρονα χρειάζεται καλύτερη στήριξη στον τομέα της γεωργίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συντονιστεί εδώ πέρα και για τις γυναίκες αγρότησες και να έχει και μια ρεαλιστική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Πέτυρ για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω τα εξής. Τι πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό η ποσότητα ή η ποιότητα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ισότητας με ένα σωρό στρατηγικές και ένα σωρό έγγραφα, εάν μας νοιάζει πραγματικά η άρση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην ποιότητα των προτάσεων, να έχουμε υλοποίηση, αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων, των υφιστάμενων μέσων που επιτρέπουν στις γυναίκες να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, να έχουν σωστές ώρες εργασίας, που, τα μέσα που καταπολεμούν τη βία εναντίον των γυναικών. Δεν πιστεύω ότι ε, η έλλειψη στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή το γεγονός ότι έχει μόνο ένα έγγραφο εργασίας, ένα non-paper είναι ε, το σωστό. Πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα και ειδικά για τις γυναίκες που έχουν οικογένειες και πρέπει να έχουν πρόσβαση στις, ε, στην αγορά εργασίας. Άλλωστε η οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια ε, έχει ανασταλεί και η οδηγία για την άδεια μητρότητας ουσιαστικά δεν βοηθάει τις εργαζόμενες μητέρες. Πρέπει ε, να κάνουμε ένα βήμα τη φορά, αλλά πρέπει να αναλύσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία και να τη βελτιώσουμε και αν, όπαξ και το κάνουμε αυτό, τότε να αρχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε νέα νομοθετήματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για την παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ. Σημερίζομαι όμως την απογοήτευση των συναδέλφων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ένα έγγραφο εργασίας και όχι τη στρατηγική. Το είπαμε και το Δεκέμβριο στην Επίτροπο Γιούροβα όταν ήρθε στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσει το έγγραφο αυτό ότι είναι ένα έγγραφο εργασίας και τίποτα περισσότερο. Σίγουρα στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις και μέσα για την επίτευξη αυτών των δράσεων και αυτά που ουσιάζουν από το έγγραφο. Είναι δύσκολο να πετύχουμε τους στόχους μας έτσι. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το εξής στο ΕΕΓΕ, το Ινστιτούτο αυτό, να εξετάσει τη δημιουργία παρατηρητηρίου για τη βία εναντίον των γυναικών. Είναι αυτό εξαιρετικά σημαντικό. Ένας Ευρωπαίος συντονιστής για την πρόληψη ε, της βίας, των περιστατικών βίας, θα μπορούσε να τεθεί επικεφαλής αυτού του παρατηρητηρίου. Τι έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη γραπτή μας δήλωση αναφορικά με το Ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών. Άνω, πάνω από 400 μέλη του Κοινοβουλίου έχουν υπογράψει αυτή τη δήλωση. Όμως προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υιοθετήσει αποφάσεις να ε, κηρύξει την επόμενη χρονιά ως το έτος για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών. Η οδηγία του 2006 για την ισότητα ευκαιριών πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν έχει αναθεωρηθεί και υπάρχουν χώρες όπου η οδηγία δεν έχει εφαρμοστεί και δεν λειτουργεί. Η συνεργασία είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό και οφείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι έχει κάνει λάθος, δεν έχει λειτουργήσει έξυπνα. Όμως υπάρχει χρόνος και μπορεί να αποκαταστήσει το λάθος της αυτό. Ευχαριστώ. κυρία Μπαρμπάρα Ματέρα, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι μέλος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και για τα Δικαιώματα των Φίλων εδώ και 7 χρόνια και τόσα χρόνια υπερασπίζομαι τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για ισότιμα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των δύο φίλων. Φέτο η Κομισιόν μα παρουσίασε ένα έγγραφο εργασία ε, που περιλαμβάνουν οι προτεραιότητέ τη η αριστερά από αυτό το κοινοβούλιο αποφασιστικά κατέκρινε τη μέθοδο εργασία τη Κορισιόν και σημειώνουμε ότι αυτό το έγγραφο δεν είναι νομικά ισχυρό. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση για δύο λόγου. Καταρχήν είμαι ρεαλίστρια που κοιτά τα αποτελέσματα που περιμένουμε και τι συγκεκριμένε λύσει για τα πραγματικά προβλήματα. Δεύτερον, το να έχουμε μία νέα στρατηγική όπου θα έχουμε μία ε, νέα νομοθεσία, ενώ έχουμε ακόμη οδηγίε που δεν έχουν εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη, δεν έχει πολύ νόημα. Το έγγραφο εργασία, ε, έτσι όπω μα το παρουσίασε η Επίτροπο Γιούροβα, περιλαμβάνει πολλέ θετικέ αναφορέ, όπω η θέληση να ενισχυθεί η καινοτομία και η δημιουργικότητα και να δοθούν κίνητρα στη γυναική επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα τη κατάρτιση και τη εκπαίδευση. Ε, έχουμε ουσιαστικά εδώ μία προσέγγιση σε ό,τι αφορά την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και εκεί βρέπουμε και ισχυρή οικονομική ενίσχυση για να προωθηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας εδώ. Ουσιαστικά τι πρέπει να κάνουμε, να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να εργαστούμε έτσι ώστε να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι γυναίκες στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ματέρα. Και τώρα η κυρία Χέντ. Από το, 2015 η Κομισιόν παρουσίασε την στρατηγική της για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Πρόκειται για ένα εσωτερικό έγγραφο εργασίας και όχι για μια επίσημη ανακοίνωση. Αυτό το έγγραφο έφερε τον τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα». Όμως έχουμε απογοητευτεί από την υποβάθμιση του εγγράφου αυτού. Η Κομισιόν απλώς ε, μας παρουσίασε ένα εσωτερικό έγγραφο στρατηγική, αλλά πρόκειται για πάτη. Εγώ θα ήθελα να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν κατόρθωσε να μας παρουσιάσει ουσιαστικά μια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων. Αν θέλει η Κομισιόν να είναι σοβαρός πρωταγωνιστής, θα την παρακαλούσα να πράξει το καθήκον της και πιστεύω ότι έχει αρκετό χρόνο για να το πράξει. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Σόγκαρ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί για τις γυναίκες, όμως ε, παρά τις νέες αυτές ε, δυνατότητες δεν έχουν γίνει πιο ενεργές οι γυναίκες στην ε, αγορά εργασίας. Είναι πολύ μικρότερη η μισθή τους, αλλά και ως προς το μέλλον τους φαίνονται φαίνεται ότι τα χρήματα δεν πρόκειται να αυξηθούν. Υπάρχουν επίσης και μεγάλες ε, διαφορές ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης, η οποία αυξάνεται. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε ε, αλλιώς για τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών, να αλλάξουμε την εικόνα που έχουμε στο κεφάλι μας. Η στρατηγική είναι στη σωστή κατεύθυνση, όμως πρέπει αυτή την κατεύθυνση να την σταθεροποιήσουμε. Ποια είναι λοιπόν η πρόθεσή σας, πώς μπορούμε να επιτύχουμε η δημιουργία οικογένειας να μην αποτελεί μειονέκτημα για τη γυναίκα και σε επίπεδο οικογένειας και μισθού και σύνταξης. Ε, ξέρετε ότι οι δημογραφικές τάσεις στην Ευρώπη δεν έχουν θετική έκβαση, θετικές επιπτώσεις, όλο και λιγότερα παιδιά γεννιούνται και γι' αυτό στα κράτη-μέλη θα πρέπει να προωθήσουμε τη δημιουργία οικογένειας μέσα από πιο ευέλικτες ώρες εργασίας. Η δυνατότητα θα πρέπει να δίνεται για κάτι τέτοιο. Οι γυναίκες δεν πρέπει να ε, είναι υποχρεωμένες να επιλέξουν ανάμεσα στην καριέρα και στην οικογένειά τους. Ευχαριστούμε πολύ ε, για τα λόγια σας και τώρα δίνω το λόγο στην κυρία Φάρν που έχει και αυτή 1,5 λεπτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους ε, για την ε, εντατική δουλειά τους να πείσουν την Κομισιό να κάνει το σωστό. Ε, δημοσίευση μιας ανακοίνωσης φιλόδοξης ε, για την ισότητα των γυναικών είναι κάτι που χρειαζόμαστε απαραίτητος. Πρέπει να είμαστε ολιστικοί και θαραλέοι, γιατί αυτό το σχέδιο θα πρέπει να διασφαλίζει ότι εσωματώνει τη διάσταση του φύλου σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τις πτυχές τους. Ας πούμε, στην πολιτική κατά της φτώχειας που είχαμε αυτό το μήνα, Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους κατά της φτώχειας έως το 2020 αν δεν έχουμε επιτύχει πραγματική ισότητα των φύλων. Η οικονομική κρίση και οι πολιτικές λιτότητας επηρέασαν τις γυναίκες δυσανάλογα. Οι ε, ανήπαντρες γυναίκες ε, βρίσκονται σε πολύ επισφαλή θέση και πρέπει να παλέψουν για να φέρουν φαΐ στο τραπέζι τους. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να κινηθεί γύρω από μια φιλοδόξη στρατηγική ω προ τα φύλλα σε όλα τα επίπεδα και πρέπει να έχουμε και ένα ευρωπαϊκό εξάμεινο που θα είναι πολύ πιο ευαίσθητο προ την ισότητα των φύλων. Πραγματικά δημονώ η ε, Κομισιόν να αναλάβει αυτή τη δράση που χρειαζόμαστε με τόσο ε, επίγοντα χαρακτήρα. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι από εσάς ε, Ήσασταν πειθαρχημένοι και τελειώσατε ε, τον, την ομιλία σας πριν το χρόνο που έπρεπε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα για 1,5 λεπτό η κυρία Μποκνιάζαν. Κύριε Πρόεδρε, η εμπειρία δείχνει ότι η στρατηγική για την ισότητα των φύλων ε, ε, δεν έχει προχωρήσει όπως έπρεπε και αυτό μας ανησυχεί. Επίσης, Υπάρχουν και άλλα σημαντικά έγγραφα που έχουν να κάνουν με την πάταξη της βίας κατά των γυναικών. Ε, το 90% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν ότι μια τέτοια στρατηγική είναι απαραίτητη. Όμως η Κομισιόν μας ε, ε, έδωσε απλώς ένα έγγραφο εργασίας και αυτό είναι κρίμα. Υπάρχουν τόσες αλλαγές στα κράτη-μέλη που πρέπει να γίνουν στην Κροατία, για παράδειγμα τη χώρα με αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει μια συζήτηση για την ε, την ε, γονιμοποίηση in vitro. Και πρέπει να συζητήσουμε πολύ περισσότερο για την ισότητα και σε άλλα επίπεδα. Ε, γι' αυτό το λόγο ζητώ από την Κομισιόν να μας οδηγήσει σε μια νέα στρατηγική για την ισότητα των φύλων, να θεσπίσει μια τέτοια νέα στρατηγική, ε, την οποία εμείς αναμένουμε με μεγάλη αδειμόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάποια πράγματα μπορεί να θεωρούνται αυτονόητα, όμως ως προς την ισότητα των δύο φύλων, θα, αντί να κάνουμε βήματα μπροστά, κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Η στρατηγική λοιπόν για την ισότητα των φύλων είναι κάτι που δεν πρέπει απλώ να το λέμε, είναι η υποχρέωσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. μισή λεπτό η κυρία Ρέγκνερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμη επίτροπε. Στην Αυστρία πολύ συχνά ε, με ρωτάνε τι μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για τις γυναίκες έχουμε τόσα επιτύχει, πραγματικά έχει ουσιαστικά αλλάξει η ζωή των γυναικών. Υπάρχουν οδηγίες, κανονισμοί, όλα αυτά είναι εξαιρετικά. Ε, τώρα όμως ξαφνικά βρισκόμαστε σε μία περίοδο φυσικασμού και ησυχίας. Τα κράτη-μέλη ε, μιλάνε για την αρχή της επικουρικότητας ε, και με αυτόν τον τρόπο φρενάρουν τις διαδικασίες. Θα πρέπει η Κομισιόν λοιπόν να μην δηλιάζει υπάρχουν προβλήματα με τις γυναίκες σε σεξουαλικό επίπεδο, σε επίπεδο υγείας. Έχουν περισσότερα προβλήματα από τους άντρες. Ε, οι γυναίκες έχουν περισσότερα προβλήματα ως προς την ανεργία, έχουν μερική απασχόληση, η ψηφιοποίηση και οι γυναίκες και οι γυναίκες και το gender budgeting. Όλα αυτά τα ζητήματα, ε, αγαπητή Επιτροπή, είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν και αυτό το έγγραφο που έχει η Κομισιόν καταθέσει ε, είναι πολύ λίγο για αυτά που χρειαζόμαστε. Είναι μια μικρή στρατηγική. Χρειαζόμαστε κάτι πιο ουσιαστικό, μια πραγματική στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Ευχαριστώ. Τώρα, τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Σάιμον, για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνεχίζοντα ε, για τόσα έλεγε η κυρία Ρέγκνερ, είπε ότι οι άνθρωποι πολλέ φορέ ε, ρωτάνε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα όταν επιστρέφω στην πατρίδα μου και λέω στους πολίτε ότι συζητήσαμε μια νέα στρατηγική τη Κομισιόν βλέπει κανεί ότι δεν πείθονται κατευθείαν ότι αυτό είναι απαραίτητο και ότι θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στη ζωή του. Όταν πας στην πατρίδα σου και του λες ότι κάνει μια συζήτηση για το γεγονό ότι η Κομισιόν δεν έχει στρατηγική Μπορεί να τους κατηγορήσεις για το ότι δείχνουν κάπως σκεπτικοί και είναι, αποδεικνύουν σκεπτικισμό για το ότι διδαπανούμε εδώ το χρόνο μας. Εκεί όπου ζω εγώ, ε, οι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια από εμά ε, εδώ, ε, γιατί δεν πρόκειται να το λάβουν από την κυβέρνησή του. Ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει αυξηθεί το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στι 4.500 λίρε το χρόνο. Είναι τεράστιο αυτό το χάσμα και ουσιαστικά οι γυναίκε έχουν πληγεί πολύ περισσότερο από του φόρου από ότι οι άνδρε και κανεί δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Στρέφονται σε εμά και σε εσά για να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Έτσι λοιπόν αυτή η μη στρατηγική που είναι αδύναμη και για τους μισθούς ε, και για την ενδοκογενειακή βία δεν είναι καλή για μας για να κάνουμε τη δουλειά μας. Πρέπει λοιπόν να πω ε, στην Επιτροπή ότι πρέπει να ανέλαβει δράση. Κύριε Σάιμον, ε, υπάρχει μία μπλε κάρτα από τον κύριο Γκερίκα. Δέχεστε. Όχι. Όχι. Αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε εδώ τον κατάλογο των ομιλητών. Δυστυχώς ε, δεν μπορούμε να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο που ζήτησε την πλακάρτα, αλλά τώρα θα δώσω το λόγο σε όλους όσους θέλουν να μιλήσουν. Παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο του ενός λεπτού. Κύριε Σόβιν. Ευχαριστώ. Οι γυναίκε έχουν κατά μέσο όρο χαμηλότερου μισθού από του άνδρε. Είμαστε πιο εκτεθειμένε στην φτώχεια όταν ε, φτάνουμε στην τρίτη ηλικία και έχουμε και περισσότερε δουλειέ στο σπίτι. Στην αγορά εργασία, πολύ συχνά βλέπουμε ότι οι γυναίκε ε, υπογράφουν σύμβαση εργασία αν υπογράψουν μια δήλωση ότι δεν πρόκειται να τεκνοποιήσουν τα επόμενα έτη. Οι γυναίκε με μικρά παιδιά επίση έχουν λιγότερε ευκαιρίε να βρουν δουλειά, επειδή μπορεί το παιδί να αρρωστήσει. Είμαστε λοιπόν σε χειρότερη θέση και στην αγορά εργασία αλλά και στην πολιτική. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Είχαμε από τις έχουμε από 25 πρόεδρους μόνο δύο γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να αναλυφθεί πολιτική δέσμευση στο υψηλότερο επίπεδο. Πρέπει να δούμε μια ανακοίνωση από την Κομισιόν για τα ίσα δικαιώματα των δύο φίλων. Δυστυχώς όμως το μόνο που λάβαμε ήταν ένα δύναμο μήνυμα. Ο πρόεδρος της Κομισιόν στέλνει ένα μήνυμα ότι δεν είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα για αυτόν. Η Κομισιόν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερο σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ, κύριο Καπούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ισότητα των δύο φύλων θα υλοποιηθεί δύσκολα χωρίς μια στρατηγική που να εξαλείφει το δομικό χαρακτήρα της ανισότητας που υπάρχει ακόμη στην κοινωνία μας. Είναι απαραίτητο η δημόσια πολιτική να μεταφραστεί σε μια συγκεκριμένη, σε ένα συγκεκριμένο έλεγχο των διαθέσιμων μέσων. Αλλά θέλουμε μια αρχή που να αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης δικαίωμα σε όλες τις συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προοπτική της ισότητας των δύο φυλών θα πρέπει να ενταχθεί σε όλες τις πολιτικές. Ήδη έχουμε αναφερθεί στην ηθική υποχρέωση να εργαστούμε προς μια ριζική αλλαγή της νοοτροπίας, ε, ε, το να καθυστερούμε, να νομοθετήσουμε. Μιλάμε ότι μας επιφέρει καθυστέρηση και δεν υπάρχει ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε παρκές επίπεδο. Έτσι λοιπόν, επιτεκτική αναγκή Κομισιόν να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική για την ισότητα των δύο φύλων. Ο κύριος Μαριάς η νέα στρατηγική της ευρωπαϊκής επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών έχει σαν στόχο την ισότητα των δύο φύλων στα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης όπου συχνά παρατηρούνται παραβιάσεις των δικαιωμάτων των γυναικών αλλά και διακρίσεις εις βάρος τους. συγκεκριμένα στον εργασιακό τομέα διαπιστώνεται ένα μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα που ανέρχεται σήμερα στο 16,4% και ένα αντίστοιχο συνταξιοδοτικό χάσμα που ανέρχεται στο. 39%. επιπλέον συχνά οι γυναίκες εργάζονται σε θέσεις μερικής απασχόλησης οι γυναίκες αποτελούν την ομάδα του πληθυσμού που έχει πληγεί περισσότερο τόσο από τη λιτότητα όσο και από τα μνημόνια. στην ελλάδα που έχει φτωχοποιηθεί από τα μνημόνια το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο οδηγεί τις γυναίκες ελεύθερες επαγγελματίες και τους αγρότες αλλά κυρίως τις αγρότισσες να διαθέτουν πλέον πάνω από το 80% του ετήσιου εισοδήματός τους για ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. γι' αυτό παλεύουν όλες αυτές οι γυναίκες μαζί με τον υπόλοιπο ελληνικό λαό ενάντια στην τρόικα και θα συμμετάσχουν αύριο στη μαζική γενική απεργία. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τερσόν. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ε, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση ε, που έχουμε και θα έπρεπε να κάνουμε και με την Επίτροπο Γιούροβα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το να θέλετε να υποβαθμίσετε μια τέτοια στρατηγική σε ένα πλόγραφο εργασία ε, δεν μα βρίσκει σύμφωνο. Έχουμε πολύ ανησυχητικά στοιχεία για την αύξηση τη ανισότητα στην Ευρώπη. Η Eurostat μα λέει ότι σε πάνω από 9 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε το χάσμα στου μισθού το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φιλόσοφων μας λέει ότι μία γυναίκα στους 25 άντρες κατέχει μία ε, ηγετικά υψηλή θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εσείς αν πιστεύετε ότι αυτό δεν αξίζει μία στρατηγική για το φύλλο, συγγνώμη, τι να σας πω, εσείς έχετε στρατηγικές όπως σε θέματα όπως η ενέργεια ε, και η θαλάσσια ασφάλεια. Αυτό το θέμα δεν αξίζει. Εγώ νομίζω ναι, σας το ζήτησε το Συμβούλιο, σας το ζητά και το Κοινοβούλιο. Σας παρακαλώ να διορθώσετε αυτό το σφάλμα και αυτή την έλλειψη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο. Νομίζω ότι η ισότητα των δύο φίλων έχει συζητηθεί επαρκώς από τους συναδέλφους. Η κυρία ε, Γιούροβα επίσης αφιέρωσε ένα ολόκληρο βράδυ για αυτό το θέμα. Ε, για, όσον αφορά τώρα την συμφωνία για τα δεδομένα και εκεί και το θέμα των γυναικών. Νομίζω λοιπόν ότι ε, όλα αυτά είναι πολύ ουσιαστικά. Βλέπουμε ότι και στην φύση τα πράγματα είναι ε, έτσι 55% γυναίκες, 45% άντρες, όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το τηρεί αυτό, αυτή την αναλογία. Υπάρχουν προκαταλήψεις κατά των γυναικών, διακρίσεις. Η ισότητα των φύλων δεν πρέπει να είναι πολιτικό φετίχα και έχω πολλές φορές την αίσθηση ότι αυτό ισχύει. Ευχαριστώ. τελευταία ομιλήτρια κυρία Τόμασιτς. Παρακαλώ καθίστε. Ευχαριστώ. Είναι λυπηρό που το 2016 ακόμα συζητάμε αυτό το θέμα παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν δώσει πολύ γενναίες μάχες ακόμα υπάρχουν διακρίσεις. Υπάρχει ευαισθητοποίηση μεν, αλλά δεν έχει επιληθεί ακόμα το ζήτημα. Το status quo που ε, ισχύει, ισχύει διότι οι μέθοδοι δεν είναι αποτελεσματικές. Τα κοινοβούλια, οι πολιτικοί ακόμα δεν έχουν βρει τρόπο για να τιμωρήσουν τις ανοιχτές διακρίσεις κατά των γυναικών. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την ε, το προνόμιο να επιβάλλουμε ποσοστώσεις ας πούμε στις ε, ιδιωτικές εταιρείες αλλά ε, δεν θα ήταν αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε θα έπρεπε να κάνουμε εκστρατείες ώστε να αλλάξουμε τις ε, νοοτροπίες της εταιρείες οι σχέσεις στις οικογένειες όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που, για τα οποία πρέπει να μαχηθούμε και πρέπει να αλλάξουμε και αυτό που πιστεύουν οι πολίτες Ευχαριστώ πολύ Τελειώσαμε με τη διαδικασία eye και τώρα δίνω το λόγο στον Επίτροπο, τον κύριο Καϊτής. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να πω. Ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ακούσω τις απόψεις σας, τις προτάσεις σας. Θα ήθελα να επενθυμίσω το εξή. Η προτεραιότητα είναι στρατηγική για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων για την περίοδο 2010-2015 παραμένει σε ισχύ. Πρέπει να προβούμε στην εφαρμογή, χρειαζόμαστε ένα πραγματικό σχέδιο δράσης, δράσης επιτόπου. Ξέρουμε ότι όλα τα κρατη έχουν τα εθνικά τους σχέδια δράσης, αλλά θα πρέπει να έχουν και τα κατάλληλα μέσα. Όλοι συμφωνούμε ότι η ισότητα των δύο φύλων σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους τους πολιτικούς τομείς και στο δικό μου χαρτοφυλάκιο και στο χαρτοφυλάκιο των συναδέλφων της κυρίας Γιούροβα. Εμείς ως Επίτροποι θα πρέπει να κατανοήσουμε με αυτόν τον τρόπο την ισότητα των φύλων να προβούμε σε δράσεις και να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε τις προτεραιότητες. Εδώ προτείνουμε στρατηγική δέσμευση για την περίοδο 2016-2019. Πρόκειται για ένα πλαίσιο αναφοράς προκειμένου να προωθήσουμε και να εφαρμόσουμε την ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα, σε τοπικό, εθνικό, και υπερεθνικό επίπεδο. Χρειαζόμαστε συντονιστικούς μηχανισμούς και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Να επαναλάβω εκ νέου. Έχουμε κάποιες δράσεις κλειδιά που πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε ένα από τους τομείς προτεραιότητας, από τους πέντε τομείς προτεραιότητας και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Και Φυσικά θα πρέπει να θέσουμε σημεία αναφοράς, χρονοδιάγραμμα και να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τις πολιτικές. Στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε καλύτερη διακυβέρνηση και πρέπει να δούμε πώς θα προβούμε στην εφαρμογή. Βλέπουμε πάρα πολλές στρατηγικές που λήγουν. Αλλά αν δούμε την εφαρμογή, υπάρχει μεγάλο κενό μεταξύ των στρατηγικών, δηλαδή μεταξύ της θεωρίας και της πράξης, την εφαρμογή στην πραγματική ζωή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας και να προβούμε σε ανταλλαγή απόψεων από την πλευρά της Επιτροπής. Εμείς θέλουμε να δούμε ενεργή βελτίωση του θέματος, δηλαδή της βελτίωσης της ισότητας των φύλων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επιτρόπε για τις τελικές σας σκέψεις. Ενημερώνω τους βουλευτές ότι αυτό είναι και το τέλος